και σχολεία. Παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Προέρχεται η προφορική ερώτηση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πρώτα-πρώτα, να δώσουμε τον λόγο στην ε, πρώτη συντάκτρια της ερωτήσεως, την κυρία Βαλενθιάνο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πρώτη μου λόγη θα ήθελα ε, να είναι το εξής. Να μπορέσουμε εμείς ως ε, Ολομέλεια να τιμήσουμε αυτή την ανεκτήμητη βοήθεια όσων δουλεύουν στις ζώνες πολέμου, δάσκαλους, νοσοκόμους, γιατρούς, όσους ε, δουλεύουν σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι οι οποίοι κινδυνεύουν με την ίδια τη ζωή τους, προσπαθούν κάτι να κάνουν για να επικρατήσει ανθρώπινη αντιμετώπιση εκεί που δεν υπάρχει πια ανθρωπιά. Οπότε θα πρέπει να γίνει συζήτηση στο Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει πολλά η διεθνής κοινότητα έχει προδώσει τον κόσμο, τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτές τις ζώνες των συγκρούσεων και μιλάμε ότι όλο ένα και αυξάνονται οι επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους όπως σε νοσοκομεία και σχολεία. Δεν νομίζω ότι κάνουμε αρκετά για να αποτρέψουν αυτές τις επιθέσεις και δεν μιλώ για μεμονωμένες περιπτώσεις. Ε, πρόκειται για μια ολόκληρη τακτική βλέπουμε να αναπτύσσεται στην Συρία και στην Ιεμένη εκεί όπου αυτές οι επιθέσεις νοσοκομεία και σχολεία ανέρχονται σε δεκάδες και τα δε σε εκατοντάδες. Αυτό ε, πλήσει χιλιάδες που πια δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και πρόκειται για εγκλήματα πολέμου. Μα και στον πόλεμο υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι σήμερα δεν τηρούνται ούτε επιβάλλονται από κανένα. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, άρα θα πρέπει να σταματήσει η ατιμορρησία. Και αντίθετα με το παρελθόν, οι άμαχοι σήμερα ε, έχουν ε, τα περισσότερα θύματα από τους πολέμους. Όλο ένα και πιο σημαντική είναι η φορήση μη κρατική σε Συρία και Ιράκ. Ε, έτσι όμως τα πράγματα μπερδεύονται στον πρώτο ανθρώπινα δικαιώματα, άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε και επίσης θα πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία τους ισχύοντες μηχανισμούς και πολλά από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι διατυπωμένα εγγράφος αλλά αυτό που θέλουμε να μάθουμε και γι' αυτό και απευθύνουμε την ερώτηση στο Συμβουλίο είναι τι έκανε το Συμβούλιο τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιν αυτή τη συστηματική καταπάτηση των δικαιωμάτων τώρα παραποτέ χρειάζεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να υπεραμείνεται των αξιών της. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό ε, αντί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σαλόμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο το οποίο δεσμεύτηκε και τήρησε την υπόσχεση να συμμετάσχει στην συζήτηση αλλά και εγώ συμφωνώ με την κυρία Βαλενθιάνο ότι θα πρέπει ε, να χαιρετήσουμε την προσπάθεια και το πόσο έτσι κάνουν τη ζωή τους όλοι αυτοί ε, οι άνθρωποι που προσπαθούν κάτι να βοηθήσουν σε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί η καταπάτηση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους αυτούς τους πολέμους Συρία, η Εμένη, η Παλαιστίνη έχουν γίνει μια καθημερινή ρουτίνα. Ε, πρόκειται για εγκληματικές πράξεις συνεχής και δεν είναι πια παράπλευρα ε, απροσδόκητα και αναπόφευκτα φαινόμενα. Πρόκειται για μια ε, στρατηγική η οποία είναι βέβαια εκούση. Επομένως έχουμε εδώ ένα πισωγύρισμα όσον αφορά τον πολιτισμό μας γιατί ήδη εδώ και 150 χρόνια άρχισαν να ισχύουν οι βασικοί, οι πρώτοι κανόνες για ανθρωπιστική συμπεριφορά σε περίπτωση πολέμου. Βέβαια τώρα έχουμε ένα σωρό κανόνες, αλλά έχουμε και ακόμα περισσότερες ε, παραβιάσεις αυτών των διεθνών κανόνων και βρισκόμαστε τώρα στο κορυφαίο σημείο ε, αναγκαιότητας του να υπάρξει ανθρωπιστική αρρωγή σε περιπτώσεις πολέμου. Ε, εκατοντάδες χιλιάδων εκτοπίζονται, γίνονται πρόσφυγες Εάν όλου αυτού βάλουμε μαζί, θα ισοδυναμούσαν με τον πληθυσμό Γαλλίας και Ισπανίας μαζί. Έχουμε πάνω από μια δεκαετία πολέμου στην Αφρική. Πέντε χρόνια τον πόλεμο στη Συρία, στην Παλαιστίνη. τέσσερι γενιές έχουν παρακολουθήσει εκεί την σύγκρουση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η ατιμορρησία και να την ανεχόμαστε. Έχουμε η ηθική υποχρέωση νομική και πολιτική να απαιτήσουμε την ε, πάυση τέτοιων επιθέσεων κατά νοσοκομείων, σχολείων, ε, τόπων λατρείας που σκοτώνουν ε, τους άμαχους, τους ανήλικους, τις γυναίκες. Η δε προφοργυρώτηση της κυρίας Βαλενθιάνο ήταν τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και εν ώψη της συνάντησης κορυφής της Κωνσταντινούπολης ζητώ από τα κράτη-μέλη δια του Συμβουλίου που τα εκπροσωπεί να δεσμευτούν ξεκάθαρα για να κάνουν κάτι ως τούτος ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο να γίνει σεβαστό μια που τόσο πολύ ο κόσμος εκεί το χρειάζεται. Ευχαριστώ κύριε Χένης Πλάσιτος, η Υπουργός. Έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ επισημαίνεται τις επιθέσεις σε βάρος ε, σχολείων, νοσοκομείων σε περιοχές συγκρούσεων. Είναι απαράδεκτο αυτό και καταδικάζουμε αυτές τις αποτροπές πράξεις. Όπως γνωρίζετε, η προαγωγή της στήρησης και του σεβασμού του ανθρωπιστικού διεθνούς δικαίου είναι καθήκον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και του Συμβουλίου ειδικότερα. Οι κατευθύνες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή της συμμόρφωσης με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο έχουν υιοθετηθεί από το 2005 και επαναβεβαιώθηκαν το 2009 από το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο πρόγραμμα δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το σχέδιο για τα 2015-2019. Στην 32η Διεθνή Διάσκεψη Ερυθρού Σταυρού και Τριχάς η διεθνη διασκεψη ερυθρου σταυρου η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίωσε τη βούλησή της να ε, υποστηρίζει πάντοτε τη συμμόρφωση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ιδιαίτερα μέσα από τις διαβουλεύσεις έκυψαν κοινά μηνύματα. Το Συμβούλιο επίσης σημείωσε στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου ότι η Σύνοδος Κορυφής για το ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις των διαφορών εμπλεκομένων μερών, διασφάλιση της ανθρωπιστικής πρόσβασης και τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κυρίως. Και ναι, βεβαίως, βεβαίως και θέλουμε να συζητηθούν οι ε, προπαρασκευαστικές εργασίες της διασκέψης του προσεχής σας σύνοδο το Μάιο. Για τα ιδιαίτερα ζητήματα μεταξύ το Συμβούλιο ε, αντιμετώπισε το θέμα της Συρίας το προηγούμενο καλοκαίρι ζητώντας από τα εμπλεκόμενα μέρη και όπως θα συνεχίσει να πράξει να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς και τις ρήψεις όλμων εις βάρος αμάχων, επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων ιδιαίτερως. Για τη Συρία το, και το Ιράκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν διατυπώσει τις ανησυχίες τους για σοβαρότατες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά σχολείων, νοσοκομιακών εγκαταστάσεων, ανοιχτών λαϊκών αγορών και το καθεξής. Το 2015 συγκεκριμένα δηλώσαμε ότι η λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων είναι σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας που, που θα επιτευχθεί και, με την, και, και εν ώψη της διαρκούς και μόνιμης λύσης του προβλήματος και θα διωχθούν όσοι είναι υπεύθυνοι για τις ε, εν προκειμένου παραβιάσεις. Ε, η συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο είναι επίσης σημαντικό κομμάτι των συμπερασμάτων για την ε, Συρία και το Ιράκ του Μαρτίου 2015. Επίσης, επί τη ευκαιρία αυτή το Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για την διασφάλιση φαρμακευτικής περιθέλεψης σε κάθε περίπτωση και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχει συζητήσει το Συμβούλιο στη συζήτηση για τη Λιβύη, για τη Λιβύη το Νότιο Σουδάν, την Ιεμένη και πολλές άλλες περιοχές ε, εμπόλεμες η προαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, προαγωγής και της απαγόρευσης των παραβιάσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων έχει και την απόφαση του 2011 της ΚΕΠΑ από το Συμβούλιο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πρέπει να εγείρουν ζητήματα συμμετοχής και παραπομπής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε κάθε συζήτηση, διαπραγμάτευση και πολιτικό διαλόγο με κράτος, ομάδα κρατών, η περιφερειακή οργάνωση ως ουσιώδες ε, μέσων για την επιβολή του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εν τέλει, παραβίασεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι ο λόγος για τον οποίο επιβάλλονται πολλά περιοριστικά μέτρα σε περιπτώσεις όπως τη Συρία τη Σιμένη του Μπουρούντι και άλλων τρίτων χωρών. Βεβαίως, και πέραν αυτών του Συμβούλιο συμμερίζεται την ανησυχία σας για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα επιθέσεις εις βάρος ε, νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αναλαμβάνει δράση αναλόγως. Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι το διεθνές δίκαιο αφορά τον άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, παιδί, οικογένεια. Και δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε, δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζουμε τη διάσταση της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς στην εξωτερική μας πολιτική. Αντιθέτως, πρόκειται για θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ <clears throat> για τα λόγια σας, για την ε, εισαγωγή αυτή για την προφορική ερώτηση. Θα έλθω τώρα στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Πρέντα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχετε τον λόγο και έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ψήφισμα που διαπραγματευτήκαμε και που συζητούμε σήμερα καταδικάζει απερίφραστα επιθέσεις κατά νοσοκομείων και άλλων μη μάχημων στόχων σε περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις. Αυτό είναι απόλυτα αντίθετο με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι η βασική αρχή του ε, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου είναι η προστασία των προσώπων που βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων. Και το κείμενο το οποίο έχει κατατεθεί είναι ισορροπημένο. Όμως η άκρα αριστερά τι κάνει, κάνει τα συνήθη, καταθέτει τροπολογίες, άσχετες με το θέμα, για τη Δυτική Σαχάρα, για την άμβλωση, για το Ισραήλ. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να αποκλίνουν με τον τρόπο αυτό από το θέμα. Ελπίζω να μην υποστηρίξουν άλλες πολιτικές δυνάμεις του αριστερού φάσματος διότι έτσι στην ουσία αποδυναμώνεται το θέμα. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει ο κ. Όπως γνωρίζουμε, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ισχύει για τις ένοπλες συγκρούσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά το κράτος δικαίου και ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο τώρα δεν υπάρχει, μακρύνεται. Έχουμε τώρα όλες ε, αυτές τις επιθέσεις κατά αμάχων ακόμα και αυτών που προσπαθούν να εφαρμόσουν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα πια σύγχυση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών στόχων και οπότε ε, αυτοί οι ουδέτεροι που προσπαθούν να ενεργήσουν έχουν γίνει στόχος. Οπότε ε, βλέπουμε ότι το προσωπικό των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων ε, θεωρούνται ως στόχος που πρέπει να πληγεί. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ε, πάρα πολλές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και επιθέσεις του στο Αφγανιστάν και αυτό γίνεται από κάποιους φορείς ή κράτη που είναι σύμμαχοι μας τον Ιανουάριο επίσης στην Ιεμένη και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε πώς στη συνάντηση κορυφής της Κωνσταντινούπολης θα αποφασιστεί επιγόντως μία ε, δράση ούτως ώστε να ε, προστατευτούν οι κινδυνεύοντες ε, φορείς ανθρωπιστικών, ανθρωπιστικής προσπάθειας και βοήθειας. Οπότε θα πρέπει να κινητοποιηθεί και το Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου. Να γίνουν έρευνες επίσης σε σχέση με αυτές τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου να αναλυφθεί δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωριστεί ότι πρόκειται για κάτι το οποίο επήγει το Συμβούλιο αλλά και είπατε εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής να δεσμευθούν ότι στην συνάντηση κορυφής θα ε, συγκροτήσουν παρατηρήσει για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Δεμές Μάκερ. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη χώρα μου, τη Φλάνδρα, όπως σε κάθε ευρωπαϊκό έθνος, με την φρικαλότητα του πολέμου. Πριν από 100 χρόνια είχαμε τη μάχη της Ιζέρ και 100 χρόνια μετά ανορθώθηκε ο πύργος με το σύνθημα ως μνημείο όχι πια πόλεμο. Και όμως 100 χρόνια μετά πόλεμος υπάρχει. Ο πόλεμος ο οποίος είναι ε, καταστροφή για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Τις ιστορίες μας τις είπαν και μας τις ξαναείπαν οι παππούδες μας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Προβάλλουν οι κάμερες τη φρικαλαιότητα του πολέμου, τους βομβαρδισμούς που δεν ε, σέβονται ούτε σχολεία ούτε νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν χώροι ασφαλής προστατευμένοι για τους άμαχους και αυτό ισχύει και για τη Συρία βέβαια, το Αφγανιστάν, την Ιεμένη, αλλά ακόμα και για την Ανατολική Ουκρανία, την οποία εγώ προσωπικώ επεσκέφθην και είδα ότι πολύ συχνά στόχοι των βομβαρδισμών είναι και τα ίδια τα σχολεία. Πρέπει λοιπόν να εγκαταλείψουμε αυτή την ιδέα της πολιτικής της υπερίσχυσης και να σταματήσουμε να θεωρούμε ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο απλώς παράπλευρη απώλεια. Πρέπει να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των βασικών αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει όμως να προσφέρουμε και, τις, και τα μέσα για την επικράτηση αυτού του ανθρωπιστικού δικαίου. Η προσεχής Σύνοδος Κορυφής για το ανθρωπιστικό δίκαιο είναι μια τεράστια ευκαιρία και πρέπει να την αδράξουμε. Κυρία Υπουργέ, γιατί οι χώρες οι οποίες το Δεκέμβριο του 2015 έλαβαν μέρος στην 32η Σύνοδο Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου του 2015, γιατί δεν επεξεργάστηκε ένα νέο μηχανισμό ώστε να εξασφαλιστεί πως θα ενισχυόταν το σύστημα του ανθρωπιστικού δικαίου. Γιατί πρέπει να επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο πάντα. Πρόεδρος Γκέρνς, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στο Κούντους, το ένα νοσοκομείο στο Αφγανιστάν βομβαρδίστηκε και έχασαν τη ζωή τους πολλοί, μεταξύ των οποίων και γιατροί χωρίς σύνορα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ε, διατύπωσε τη λύπη τη για την καταστροφή αυτή, υπογραμμίζοντας πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Μας ε, συγκλονίζει το γεγονός ότι τα δεδομένα του GPS της ε, γεωγραφική θέση του νοσοκομείου αυτού ήταν γνωστά στι ε, αμερικανικέ αρχέ που ήταν υπεύθυνε για τον βομβαρδισμό. Δεν του εμπόδιζε όμω αυτό ε, να προχωρήσουν στον βομβαρδισμό και να οδηγήσουν στο θάνατο πολλά, πολλούς ασθενείς και ιατρικό προσωπικό. Η προσεχή σύνοδο λοιπόν ε, για την επιβολή του ανθρωπιστικού δικαίου τη Κωνσταντινούπολο πρέπει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό και την ε, ακεραιότητα των ε, εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα που πολλές φορές ε, θυσιάζουν χρόνο, ενέργεια και γενεοδορία για να δώσουν ανθρωπιστικές λύσεις. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε λύσεις τόσο προληπτικές όσο και ενδεχομένως αποτρεπτικές εν ώψη των πολυάριθμων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μεταξύ αυτών, απαγόρευση πώληση όπλων στους εμπλεκομένους φορείς ή σε εκείνους που ενδεχομένως να εμπλέκονται σε παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου. Υπογραμμίζουμε επίσης την δέσμευση για ανεξάρτητη διερεύνηση και παραπομπή για τα εγκλήματα αυτά, διεθνού χαρακτήρα, περιλαμβανομένου και του διεθνού Πενικού Δικαστηρίου. Εάν μπορέσουμε να θέσουμε ένα τέρμα στην ατιμορρησία, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και το κύριο των ΗΠΑ ω οργανισμού υπεύθυνου για τη διαχείριση των συγκρούσεων, των ένοπλων συγκρούσεων. Και θα ήθελα ιδιαίτερω να επιμείνω ω προ την ε, αδύρυτη ανάγκη τα κράτη-μέλη να τιμήσουν επιτέλου τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Κονέτσνα. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια του περασμένου Οκτωβρίου η ομάδα μου της Ενωτικής Αριστεράς ανέλαβε την πρωτοβουλία να περιλάβει ένα έξτρα θέμα στη μέση διάταξη μετά από την επίθεση του Αμερικανικού στρατού στο νοσοκομείο των γιατρών χωρίς σύνορα στο κουντούζ του Αφγανιστάν. Όλοι τότε είχαμε εκφράσει τη λύπη μας για το τραγικό γεγονός. Τι έγινε έκτοτε, οι Αμερικανοί διεξήγαγαν εσωτερικό έλεγχο, έρευνα και το σκάνδαλο έσβησε σιγά σιγά όπως οι φωνές άλλωστε των ασθενών και των γιατρών που έχασαν τη ζωή τους στο νοσοκομείο αυτό. Η ε, Διεθνής Επιτροπή στην βάση του μηχανισμού ε, εξέτασης που έχει ξεκινήσει από το 1991 με ιδιαίτερο πρωτόκολλο τη Σύμβαση τη Γενέβη και που ποτέ δεν έχει χρησιμοποιηθεί ωστόσο ως τώρα. Ιδρύθηκε λοιπόν ε, η Επιτροπή αυτή. Όμως δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή τα συμβαλόμενα μέρη στη συνθήκη αυτή, στη σύμβαση συγγνώμη αυτή. Όμως οφείλουμε επιτέλους να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αντιμετωπίσουμε το γεγονός αυτό. Καταστρέφονται νοσοκομεία από πολεμικές επιθέσεις. Αν δεν δείξουμε τους πραγματικούς υπεύθυνους θα συνεχίσουν τα πράγματα αυτά όπως έγινε και στο Αφγανιστάν και στην Ιεμένη και στην Συρία. Δεν με ικανοποιεί η απάντηση του Συμβουλίου ότι παρακολουθεί την κατάσταση και λαμβάνει μέτρα. Θέλω μια πραγματική λύση. Διότι μόνο αν κατατρομάξουμε τους επιτιθέμενους μπορούμε να αποφύγουμε επανάληψη των ε, επιθέσεων αυτών. Η κυρία Λόχμπιλερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πραγματικά λυπηρό ότι οι χώρες μέλη γίνονται συνένοχοι βαριών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Χώρες οι οποίες λαμβάνουν οπλισμό από χώρες μέλη της Ένωσης είναι υπεύθυνε εν τέλει για επιθέσεις κατά αμάχων μεταξύ αυτών και βομβαρδισμών σχολείων και νοσοκομείων. Στο προκείμενο ψήφισμα ζητούμε αποτελεσματικά μέτρα για να πάυσει η συνενοχή αυτή και ζητούμε να υποστηριχθεί η πρόταση των πράσινων για επιβολή εμπάργο εξοπλισμών από την Ευρώπη απέναντι σε τέτοιες χώρες. Το ψήφισμα αυτό βασίζεται σε προηγούμενη έκκλησή μας για την επιβολή εμπάργου εξοπλισμών στη Σαουδική Αραβία λόγω της εξτατείας της στην Ιεμένη. Οι κατευθυντήρες γραμμές για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωση προβλέπουν και άλλα μέτρα. Εμείς όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πράττουμε αρκετά για την εφαρμογή τους. Περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά και την υποστήριξη αποστολών για συγκέντρωση στοιχείων για ε, εγκλήματα πολέμου και για την υπαγωγή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Για να γίνει η δίωξη αυτά είναι αναγκαία, για να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους υπευθύνους και για να αποφευθούν μελλοντικέ θανατώσεις αμάχων. Όλο και περισσότερα σχολεία και νοσοκομεία δέχονται επιθέσεις και αυτό είναι μαρτυρία αδιάψευτη της ε, διάβρωσης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Είναι αναγκαίο, ουσιώδες, να παραμείνουν προστατευμένα σχολεία και νοσοκομεία. Η επικείμενη διάσκεψη κορυφής για το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο θα μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για να τονιστεί για άλλη μια φορά η ανάγκη συμμόρφωσης με τις αρχές του δικαίου αυτού και να βελτιωθεί η κατάσταση γυναικών νεαρών κοριτσιών και άλλων ευάλωτων ομάδων που εμπλέκονται σε πολεμικές σειράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, απαντάει η Πρόεδρος. Ο κύριος Καστάλντο, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το να γίνονται στόχοι τα σχολεία και τα νοσοκομεία απαγορεύεται ρητός από τους κανόνες του Διεθνούς και Δικαίου και ο τους είναι έγκλημα πολέμου παρ' όλα αυτά. Η διεθνή κοινότητα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μάρτυρα πολλών τέτοιων φρικτών επιθέσεων όπω του γιατρού χωρί σύνορα, τα νοσοκομεία στο Αφγανιστάν, στην Εμένη ή την Συρία, οπότε θα πρέπει ε, να συγχαρηρούμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις για το θάρρος τους. Οπότε χρειάζεται άμεσα δράση αποφασιστική, ούτως ώστε να αποκρούσουμε αυτά τα εγκλήματα και να σταματήσει φυσικά η ροή των όπλων προς τους εμπολέμους. Έκλεισε προς την κυρία Μογκερίνη, ούτως ώστε να αναλάβει πρωτοβουλία και έτσι να επιβληθεί εμπάργκο όπλων προς τα κράτη τα οποία παραβιάζουν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Να σταματήσει η πώληση των όπλων. Αυτό είναι παραβίαση του τόσο αποφάσισε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου. Ε, δεν θα πρέπει να είμαστε συνένοχοι με τη σιωπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των ομιλητών εκ μέρους των ομάδων και παρακαλώ τον κύριο Ζαμπόρσκα να λάβει το λόγο. Κύριε Ζαμπόρσκα. Πρόεδρε, Βλέπουμε δυστυχώς μια τάση να βομβαρδίζονται σχολεία, νοσοκομεία. Η τάση ήταν να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Έχει ένα καθήκον το σχολείο, όπως και το νοσοκομείο, να προσφέρει βοήθεια στον άμαχο, στον άνθρωπο, και είναι έγκλημα το να ε, επιτίθεται κανείς κατά σχολείων και, και νοσοκομείων. Λυπούμε ιδιαίτερως που κατέθεσαν προτάσεις τροπολογιών οι συνάδελφοι της ΓΚΟΕ. Γιατί έτσι βλέπω πως συμπεριφέρονται κατά τρόπο ανεύθυνο και θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ζαμπόρσκα. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Βάτενχολτσερ. Δύο Εγκλήματα πολέμου ή τρομοκρατικές επιθέσεις είτε από κρατικούς φορείς είτε από άλλους βρίσκονται δυστυχώς πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Βλέπε Συρία, Ιράκ και αλλού. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι βέβαια οι επιθέσεις κατά νοσοκομείων, σχολείων και παιδικών σταθμών πρόκειται για μια κοινική μορφή βίας, το ίδιο όπως και επιθέσεις κατά μη κρατικών οργανώσεων και όλων των άλλων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου και οφείλουν να αχθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως αυτή η πεποίθηση σε τι να βοηθήσει τους θυγωμένους. Γι' αυτό το ψήφισμά μας είναι σημαντικό. Υπενθυμίζω ότι Έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο, τις κατευθυντικές γραμμές του 2009 για, το διεθνές, για την αντιμετώπιση από πλευράς διεθνούς δικαίου τέτοιων περιπτώσεων. Θα πρέπει το Συμβούλιο να μας διευκρινίσει ποια μέτρα ελήφθησαν στο χρονικό αυτό διάστημα για να γίνουν δεσμευτικές οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές. Γνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ενώσης και των χωρών μελών Τονίζουμε τη σημασία του περιεχομένου του ψηφίσματος, τη συνεργασία που είναι αναγκαία και στα πλαίσια των Ενωμένων Εθνών και μεταξύ των χωρών μελών της Ένωσης. Ε, μια σημαντική πτυχή, ωστόσο, δεν θα πρέπει να λησμονηθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την Ιεμένη προ λίγων εβδομάδων τόνισε ξανά και νομίζω ότι δικαίως το επαναλαμβάνουμε εδώ ότι θα πρέπει να αποκλειστούν χώρες από, από ε, αποστολές εξοπλισμών που παραβιάζουν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε επιθέσεις πανταχώθεν. Έχουμε επιθέσεις και στο Άντεν. Στοχευμένη επίθεση αυτή. Κατά νοσηλευτριών που φωνεύτηκαν νοσηλεύτες, φωνεύτηκαν και ασθενείς. Η ατζέντα μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλουσιότατη. Δυστυχώς κάπου δεν το προσέξαμε το γεγονός αυτό, την επίθεση αυτή που αναφέρω στο Άντεν. Κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοια γεγονότα όπου αθώοι άμαχοι πέφτουν θύματα επιθέσεων και φωνεύονται πρέπει να τα συζητούμε και στην περίπτωση αυτή επαναβάλλεται μια στοχευμένη επίθεση Ευχαριστώ Κυρία Σάντσα, για ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε σε αυτή τη ε, στιγμή ο Γενικός Γραμματείας του χτύπησε το καμπανάκι όσον αφορά τη συνεχή του των κανόνων του Διεθνού Ανθρωπιστικού Δικαίου. Οπότε τώρα ήρθε στην ώρα το αυτό το ψήφισμα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ απογοητευτικό να βλέπουμε ότι τα περισσότερε πολιτικέ ομάδε ε, ε δεν λένε ε, τίποτα για την Δυτική Σαχάρα και για την Παλαιστίνη ε, γιατί και εκεί ισχύει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο οπότε εκεί έχουμε χιλιάδες αμάχων οι οποίοι πλήσονται σε αυτά τα κατεχόμενα εδάφη αυτή είναι αβοήθητη ε, θα πρέπει να δούμε τι είπαν για δουλειά της Γάτζας οι ερευνητικές επιτροπές το 2014 μιλούσαν για εγκλήματα πολέμου με τα νοσοκομεία που βομβάρδιζαν και για τη δυσανάλογη χρήση ισχύω και βίας οπότε θα πρέπει να ισχύσει το Εθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο οπότε τελικά για πολιτικούς λόγους δεν εφαρμόζεται το Εθνές Δίκαιο και υπάρχει ατιμορρησία ελπίζουμε αύριο να ψηφίσετε τις τροπολογίες που κατεβάσαμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Στήρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, μόνο το Φεβρουάριο του 2016 είχαμε παραπάνω από ε, χίλιες επιθέσεις κατά παρόμοιων ε, ε, φορεών στην Συρία συνήθως από τον στρατό του Άσαντ άμαχοι, νοσηλεύτριες, άλλα πρόσωπα που εργάζονται στους φορείς αυτούς έπεσαν θύματα. Δεν υπάρχει πλέον το αναγκαίο προσωπικό για να βοηθήσει τους αμάχους. Η προσπάθεια που κάνουν τα πρόσωπα αυτά είναι αξιοθαύμαστη επιθέσεις κατά νοσοκομείων αποτελούν βαρύτατη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Δεν αρκεί να τις καταδικάζουμε. Πρέπει να δράσουμε και πρέπει να αχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της διεθνούς ποινική δικαιοσύνης. Γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι επιθέσεις αυτές. Όπως για παράδειγμα και ε, ακόμα τα υποκείμενα εκείνα που κατά διαταγές του Μιλόσεβιτς επιτέθηκαν και ακόμα παραμένουν ατιμόρυτοι. Κύριε Απόστο, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ένα νέο είδος πολέμου. Επιθέσεις κατά παιδιών, γυναικών, αμάχων. κατά των κτηρίων στα οποία βρίσκονται. Πρόκειται για ένα νέο είδος πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρκεστεί λοιπόν στο να καταδικάζει, γιατί θα διέπρατε η ίδια έγκλημα αν το έπρεπε αυτό. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν δευτερείς γραμμές, πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπέτη και αν παραμείνουμε αδρανείς σε αυτής της κατάστασης θα δούμε ακόμη περισσότερες επιθέσεις και νεκρούς. Το Συμβούλιο πρέπει να προτείνει απαγόρευση ε, εξοπλισμών στις χώρες που διαπράττουν αυτά τα έγκληματα. Η συνέχιση των πωλήσεων όπλων προς τις χώρες αυτές συνιστά παραβίαση του εθνούς δικαίου. Είναι ενισχυτικό ο αριθμό των ε, θυμάτων και πρέπει να αναπτύξουμε μια κοινή θέση στο πλαίσιο του παγκόσμιου εφοπλισμού που πρέπει να είναι ο στόχο όλων μα. Η Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμασιτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η παραβιάση του Διεθνού Ανθρωπιστικού Δικαίου όπως αυτές ε, οι επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων πρέπει να καταδικαστούν τα... οι πέτοι αυτών των επιθέσεων πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη μια τέτοια συμπεριφορά δεν μπορεί για κανένα στρατηγικό λόγο ή συμφέρον να, γίνει, να θεωρηθεί ανοιχτή επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω το, το νοσοκομείο του Μπούκοβαρ κατά τον πόλεμο στην Κροατία κατά την ε, πολιορκία του Μπούκοβαρ είχε δεχθεί πολυάριθμες επιθέσεις στο νοσοκομείο αυτό και οι τρομοκράτες όταν έπεσε η πόλη ε, μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο, πήραν ε, ομήρους τους ασθενείς από τα κρεβάτια τους και το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό και τους εκτέλεσαν. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμα επιστραφεί από τη Σερβία τα έγγραφα τα σχετικά με το νοσοκομείο και οι πληροφορίες και δεν έχουν διατεθεί πληροφορίες σχετικά με τη μοίρα των θυμάτων αυτής της επίθεσης. και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σε αυτό υποστηρίζουν τη Σερβία και ε, καταδικάζουν την Κροατία η οποία δεν δέχεται αυτόν τον εξευθερισμό. Ο κύριος Χόιτ. Δεν ε, μπορούμε να αρνηθούμε το φαινόμενο των 358 διαφορετικών επιθέσεων από το 2011 και μόνο στη Συρία κατά νοσοκομείων και ε, σχολείων με την τελευταία αυτή που αναφέρθηκε στο Αφγανιστάν το νοσοκομείο των γιατρών χωρίς σύνορα και την Ιεμένη. 610 γιατροί οι οποίοι έχουν χάσει με βάση τις ε, πληροφορίες των εθνών οργανώσεων ε, μέσα σε ένα χρόνο τη ζωή τους από τις επιθέσεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο σε Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσουμε την, νόμιμη, την ένομη προστασία που θα θα παρέχεται σε διεθνέ επίπεδο, πρέπει να επιμείνουμε ώστε τα κράτη-μέλη με κανέναν τρόπο να μην ανέχονται έστω και σιωπηρά αυτέ τι επιθέσει. Πρέπει να πατάξουμε του τρομοκράτε και αυτέ τι ένοπλε ομάδε οι οποίε χρησιμοποιούν του αμάχου ω ανθρώπινη ασπίδα. Τα θύματα της βία καταφεύγουν στα νοσοκομεία για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, για να θεραπευτούν, να κλείσουν τα τραύματά τους και η τραγική ηρωνία είναι ότι μέσα στα νοσοκομεία αυτά πέφτουν ε, θύματα επιθέσεων. Εμείς καταδικάζουμε το ίσις γιατί επιτίθεται κατά των νοσοκομείων και αν θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από αυτούς πρέπει να μην παραλάβουμε το ίδιο λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ολοκλώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών ε, ε, και περνάμε στο Catch the Έχετε όλοι από, από ένα λεπτό. Κύριος Πόλτσακ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για αυτά που ο κ. Χάουιτ μόλι λίγο πριν από μένα. Υπάρχουν πολλέ τέτοιε επιθέσει. Εγώ επιθυμώ ωστόσο να ε, επικεντρωθούμε και σε άλλε, όχι μόνο σε επιθέσει που έγιναν στην Καμπούλ. Και όλε οι επιθέσει που έγιναν πέρσι στι 15 Φεβρουαρίου Φωνεύθηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση 50 άνθρωποι. Άλλοι στο Σαμίν αργότερα. Εκφράζω τη λύπη μου για όλα αυτά τα θύματα αεροπορικών επιδρομών που όντως παραβιάζουν διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Εν ώψη του ψηφίσματος της ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς, ωστόσο πρέπει να είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί, διότι είναι μονομερής η διατύπωσή της. Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη έκθεση όπως ήταν η αρχική πρόταση και όχι όπως αυτή που εμφανίζεται τροποποιημένη από την Ερωτική Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τους τελευταίους μήνες δυστυχώς έχουμε επανειλημμένα συζητήσει τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στα πεδία του πολέμου, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω της δράσης των τζιχαντιστών του ΝΤΑΕΣ όμως τον περασμένο νοέμβριο οι ηνωμένες πολιτείες ομολόγησαν τον δολοφονικό βομβαρδισμό νοσοκομείου των γιατρών χωρίς σύνορα στο αφγανιστάν. στην ιεμένη η αραβική συμμαχία της οποίας ηγείται η σαουδική αραβία έχει επιτελέσει ένα όργιο βιοαπραγιών κατά του αμάχου πληθυσμού με πολλές επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία. με τη στάση δύο μέτρα και δύο σταθμά που υιοθετεί σήμερα η ευρωπαϊκή ένωση και η δύση ευρύτερα διακυβεύεται η υπόλοιψη και η αξιοπιστία τους οι διεθνεί οργανισμοί έχουν καθήκον να αναγνωρίσουν τα εγκλήματα πολέμου στην ιεμένη το αφγανιστάν στο ιράκ και στη συρία αλλά και αλλού από όποιου και αν τελούνται. αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα ώστε οι ηθήνοντες να αναλάβουν τι ευθύνε των πράξεών του, την οικονομική αποκατάσταση των ζημιοθέντων χωρών και των ανθρώπων αλλά και την ασφαλή και ανεφόρον περίθαλψη των χιλιάδων προσφύγων που έχουν δημιουργήσει. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Έχετε το λόγο κύριε. Λίγα φαίνεται μάθαμε από τα όσα συνέβησαν από, στον, στον πόλεμο μάλλον της, ε, ε, στην επικράτεια της πρώην Ιουγκοσλαβίας σχολεία θυσίες αποτέλεσαν στόχους επιθέσεων πριν από 20 χρόνια. Θυμηθείτε το νοσοκομείο του Βούκοβαρ. Μου φαίνεται όμως ότι τελικώς τίποτα δεν διδαχτήκαμε. Πώς μπορούμε να εμφανιζόμαστε έκπληκτοι βλέποντας αμάχους να γίνονται θύματα πολεμικών επιθέσεων. Σε κάθε πόλεμο τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να διεξάγεται η συζήτηση αυτή χωρίς να συνεπάγεται σαφείς αποφάσεις αυστηρότητα της καταδίκης αυτών των βαρύτατων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κύριος Λούκας, ευχαριστώ. Συμφωνούμε με τις γενικές αρχές από τις οποίες πηγάζει αυτή η συζήτηση, αλλά βέβαια θα πρέπει να αναφερθούμε και στις αληθείς αιτίες αυτών των συγκρούσεων. Ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ΝΑΔΟ, τον είπα, για τα όσα είναι στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ευθύνη της Δύση και των συμμάχων της. Αυτοί ευθύνονται για τις επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων. Πρόκειται για εγκληματικέ ενέργειες και το Ισραήλ επίσης έχει βομβαρδίσει παιδιά ε, η Σαουδική Αραβία ευθύνεται για όσο είναι στην Ιεμένη και με τα μη επανδρομένα αεροπλάνα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έτσι καταπατούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τώρα ο Υπουργός η κυρία Χένης Πλάσκατα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλα τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου των αρχών του και των διαταξιών του είναι ε, το πνεύμα που διαπνέει την εξωτερική μας δράση. Και όπως προείπαμε απόψε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην απαρνηθούμε τις θεμελιώδεις αξίες που στηρίζουν το διεθνές δίκαιο ε, τους ανήλικους αλλά και ενήλικους. Οπότε ως προς την ε, κυρία, τον κύριο Ντεμές Μάγκερ θα πρέπει να πω ότι και εγώ όπως και εσείς καταδικάζω το ότι δεν βρέθηκε ένας μηχανισμός αποτελεσματικός μέχρι σήμερα αλλά ξέρετε τα 28 ε, κράτη-μέλη, τα περισσότερα έχουν συμμετάσχει στην ε, διάσκεψη που έγινε. Και είχαμε τη διάσκεψη αυτή του Ερυθρού Σταυρού, στην οποία αναφερθήκατε και ήδη είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε την δεσμευσή της για να υποστηρίξει το Εθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Και η Ένωση και τα κράτη-μέλη τοποθετήθηκαν και κατά της επίθεσης ε, εναντίον των γιατρών και των ασθενών. Τα κράτη-μέλη έχουν ισχυρή φωνή εάν είναι ενωμένα. Αλλά θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν ε, και όχι ορισμένα μόνο όπως έγινε στην περίπτωση εκείνης της διάσκεψης. Η Πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώνεται ε, αυτό το σημείο της διάταξης.